Ε, για να μπορέσει να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη αυτό το ψήφισμα, πράγμα το οποίο θα γίνει ε, σε συνδυασμό με τη συνάντηση του ΟΗΕ με την ε, Αφρικανική Ένωση. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω καθώς και τους ανώτερού σας, κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου, διότι βοηθάτε την Επιτροπή μας και βοηθάτε και τη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ιδίως για ό,τι είπατε για την αποτελεσματικότητα και την ε, συνέπεια. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σίνκλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συγχαίρω την εκπρόσωπο της Σουηδικής ε, Κυβέρνησης για την παρουσίασή της. Έχει μεγάλη παράδοση στον τομέα αυτό η Σουηδία, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά έχουν μεγάλη σημασία τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίω στις δικές μας χώρες. Τι κάνει η Σουηδία για να διασφαλίσει ότι κάποιες από τα νεότερα μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Και τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνόησε τη βούληση των ε, πολιτών της Ιρλανδίας και την αρνητική τους ψήφο στο δημοψήφισμα πέρυσι. Θα έπρεπε, λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναμεχθεί σε αυτή τη διαδικασία δημοψηφίσματος και δεν θα προσπαθήσει να εκφοβήσει ούτε να επηρεάσει την ε, τοποθέτηση των Ιρλανδών πολιτών αυτή τη φορά σε αυτό το δημοψήφισμα. Ευχαριστούμε κύριε Συγκλέρο. Κύριε Σόουιτ. Πρόεδρε, και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Χάμερ για την ε, παρουσίασή της και συνολικά για το πρόγραμμα της Σουηδικής Προεδρίας. Έχουμε ψηλές προσδοκίες τώρα από την Προεδρία σας. Και ελπίζω ότι στο τέλο του διαστήματο αυτού θα έχουμε την ευκαιρία να σα δώσουμε περισσότερα συγχαρητήρια παρά να σα κάνουμε επικριτικά σχόλια. Για τον κύριο Μπιόλ να ευχαριστήσω για τον συνεχιζόμενο αγώνα του ε, εισηγητού για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπόθηκαν πολλά. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθώ και εγώ σε λίγα ζητήματα. Να εκφράσω την στήριξή μου για τι δεσμεύσει σε σχέση με την ε, με τους προσώπους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ζητήματα των αποστολών ε, SDP και την εκπαίδευση σε σχέση με τα ζητήματα φύλου, τα δικαιώματα των ε, διαφορετικών ε, ομάδων σεξουαλικών προτιμήσεων που θα έπρεπε να γίνονται σεβαστά τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των ε, ιδιαίτερων μηχανισμών και των μηχανισμών συγκεκριμένων χωρών και να έρθω τώρα και στα ερωτήματά μου. Το Κοινοβούλιο στήριξε την διαδικασία mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σημαντικό εδώ είναι να θυμίσουμε ότι πολλά απομένουν να γίνουν να δούμε τι γίνεται στις χώρες μας και γιατί κάποιες φορές εργαζόμαστε ξεχωριστά σε σχέση με άλλες ε, μεταξύ χωρών αλλά και σε σχέση με το τι κάνει το κάθε θεσμικό όργανο ή οι ομάδες του Συμβουλίου μεταξύ τους. Και ως προς τις πολιτικές μας δηλώσεις, τα λόγια που χρησιμοποιούμε πρέπει να υπάρξει mainstreaming για κρίσιμα ζητήματα, καθοριστικά ζητήματα και αποφάσεις που λαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να την χάνουν τις προσοχές που τους αξίζει στην απάντησή σας, ίσως να μας δώσετε και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς προτίθεστε να κάνετε κάτι στην πράξη για όλα αυτά, γιατί τα λόγια είναι πιο εύκολα από τα έργα και ο τομέας της εμπορικής μας πολιτικής εκεί δεν είμαι βέβαιος ότι αναφέρουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες συμφωνίες που πρέπει να συζητηθούν όπως την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με χώρες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά, για να μην πω ότι βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση. Έπειτα, ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες. Εδώ στηρίζω την ε, δέσμευση όμως κάποια κάτι μέλη προτίθενται να εκφράσουν επιφυλάξεις και εμείς θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των επιφυλάξεων αυτών. Ποιες είναι λοιπόν οι δικές σας προθέσεις ως προς το θέμα αυτό. Επίσης εκφράζω τη στήριξή μου για την πρωτοβουλία σας για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ελπίζω εδώ να έχει ανάμειξη και το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, μας έχει απασχολήσει το ζήτημα αυτό και θα συνεργαστούμε με την Προεδρία σας. Απλώς να επισημάνω ότι για μένα ως πρώην ε, συγητή για το ζήτημα αυτό στο Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο όπως ο καθηγητής Ρέικη προτείνει το ζήτημα να ενισχύσουμε την προσέγγιση αυτή, αλλά να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και στο τέλος της, Ευρω... της χρονιάς θα δούμε τι κάναμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υλοποιήσουμε όλες τις υποχρεώσεις που προέκυψαν εδώ ή ίσως να θέσουμε πλέον λιγότερο φιλόδοξους στόχους. Αυτό είναι ένα ερώτημα λοιπόν που μπορώ να σας θέσω. Και κατά τέταρτον, το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και πώς το αντιμετωπίζουμε είναι κρίσιμη σημασία, νομίζω περισσότερο από πολλά άλλα, και το Συμβούλιο Ανθρώπινης, ε, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συνεχίζει να ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά να χάνει και την αξιοπιστία του. Θα πρέπει λοιπόν εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αγωνιστούμε ενάντια τη κατάσταση αυτή, προσπαθώντα να βρούμε τρόπου να καταλήξουμε σε θέσεις συνένεσης για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Ελπίζω ότι αυτό θα απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά και ιδίω την Προεδρία σα. Και τέλο, ένα προσωπικό μια προσωπική ευχαριστία για την πρόσκλησή σας προς τον πρόεδρό μας, προς τον πρόεδρό μας να συμμετάσχει στα, συζητήσεις σας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να προτείνετε ε, να τίνετε τέτοια χείρα συνεργασίας προς το Κοινοβουλίο μας και στο έργο σας στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα συνεχίσετε να συνεργάζεστε με το Κοινοβούλιο σε οπέδο θεσμικό. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θέμα τη Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, γιατί εκεί λογικά θα γίνει συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρατε και εσεί στην παρουσίασή σα. Έχει αλλάξει όμως το χρονοδιάγραμμα της ε, συνόδου αυτή και η προετοιμασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα εν του Συμβουλίου θα έχει αλλάξει τότε. Πρέπει λοιπόν να τα ξαναδούμε όλα αυτά και να συνεννοηθούμε. Ελπίζω ότι θα το συζητήσουμε και αυτό, διότι η Ολομέλεια του Δεκεμβρίου για το Κοινοβούλιο έχει γίνει πραγματικά μια Ολομέλεια που θα επικεντρωθεί στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος ίσως επηρεάσει τα πράγματα. Να το δούμε λοιπόν αυτό και να είμαστε βέβαιοι ότι η προβολή που επιδιώκουμε θα επιτευχθεί. Και να σας επιθυμίσω τις ε, συνεχείς ε, συστάσεις του Κοινοβουλίου μεταξύ των οποίων μία λέει ότι πέραν των εμπορικών μας προτεραιοτήτων πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην ε, εμπιστευτική προσέγγιση της Προεδρίας. Η ιδέα σας λοιπόν να προχωρήσετε με διαφάνεια είναι πολύ καλή. Ελπίζουμε αυτή η συγκεκριμένη σύσταση του κυρίου Μπιόλ στην αυξημένη σα αυτή η πρόθεση να δράσετε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ληφθεί υπόψη. Και ο διαθεμένος διάλογος για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Δημοκρατία είναι ελπίζω κάτι που θα εξακολουθήσει. Ελπίζω επίση ότι θα συμφωνήσουμε και για το σχετικό μηχανισμό και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή για το στόχο αυτό και τα προγράμματα εκδημοκρατισμού της Επιτροπής ε, θα οδηγηθούν σε αίσιο πέρας. Τέλος, και με συγχωρείτε που έχω τόσο πολλά ερωτήματα, Πρόεδρε. Ναι. Ο κ. Ε, Μάρτινος συνάδελφος, έπρεπε να φύγει, αλλά ζήτησε εκ μέρους του να θέσω ένα ερώτημα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν η Προεδρία σας πρόκειται να συζητήσει, να τοποθετηθεί σε σχέση με την επιστροφή του κ. Μικιάκη από την Σκοτία. Έχει κάποια άποψη η Προεδρία σας για το θέμα αυτό. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Και θα επηρεάζει τις σχέσεις Λιβύης ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Ίσως και τις Ευρωπαϊκές Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι διεθνούς, ε, διεθνούς το το ζήτημα και επειδή είναι σοβαρό, ελπίζω να θέλετε και εσείς να το συζητήσουμε. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε να το απαντήσετε κι αυτό. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Έχω ακόμα συναδέλφους που ζητούν το λόγο, ξέρετε. Και είναι σημαντικό αυτό, αλλά θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε σε αυτά. Κλείνει ο κατάλογος. Διαβάζω τα ονόματα και θα σας δώσω μέσα το λόγο για να προχωρήσουμε και στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Κιόνκα, εκπρόσωπο του κυρίου Σολάνα. Παρακαλώ, κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τη Σουηδική Προεδρία. Το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο και η πολιτική βούληση ε, πραγματικά πολύ μεγάλη. Εγώ είχα το προνόμιο να συνεργαστώ ε, με τις Σουηδικές Αρχές και δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή ότι προτίσετε να υλοποιήσει όλα αυτά που μας είπε. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, πολλά τα εμπόδια και τα περιθώρια ελιγμών ε, άκρος περιορισμένα πολλές φορές. Ορισμένοι επίσης διέπονται από τις επιταγές της Real Politik, όπως τα αποκαλούν αυτά. Δηλαδή υπάρχουν κυβερνήσεις ε, που δεν σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα και διαπραγματεύονται αυτά τα θέματα μαζί μας και κλεισμάτων των θυρών για να μην θίξουμε και τίποτα business που γίνονται εκεί. Και ε, οι προκάτοχοί σας έσπασαν τα μούτρα τους, να το πω έτσι, γιατί προσπάθησαν να εγγράψουν ε, στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κάποια θέματα να θίξουν κάποιες κυβερνήσεις για το πώς συμπεριφέρονται και πώς ασκούν την ανησυχία τους στον ΟΗΕ. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Και επίση γνωρίζουμε πόσο περίπλοκες είναι οι σημερινές ε, σειράξεις. Ε, θέλω να σας πω το εξή Πριν από λίγα χρόνια και μετά από έτοιμα του ΟΗΕ, συστάθηκε ένα πάνελ πενταμελές ε, και εκεί συμμετείχε και η χείρα του κυρίου Πάλμε ε, και έγραψαν ένα βιβλίο για τη Ρουάντα με τίτλο «Η γενοκτονία που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει». Πολύ αργά βέβαια ήρθε αυτή η μελέτη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το βιβλίο και τουλάχιστον έβαλε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και ε, κατέδειξε ε, ευθύνε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω το εξής και σας παρακαλώ να δεσμευτείτε γι' αυτό εξ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτημα. Εδώ και λίγες μέρες μας έχουν ζαλίσει με το υποτιθέμενο τέλος του πολέμου στον Ταρφούρ. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σταματούν ε, και οι βιασμοί των γυναικών που το βράδυ πηγαίνουν να βρουν νερό. Ή τελειώσαν οι βομβαρδισμοί, δεν έχουμε τίποτα να βομβαρδίσουμε και σταμάτησε ε, ο πόλεμος. Γιατί είναι σε τεχνική ανεργία που δεν έχουν τίποτα να βομβαρδίσουν τα βομβαρδιστικά αλλά δεν έχει έρθει η ώρα των ευθυνών. Και ζητώ λοιπόν από τη Σουηδική Προεδρία να δεσμευτεί ρητά και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταρτιστεί η μελέτη για τις πραγματικές ευθύνες. Για το τι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, το ποιο τελικά έφτεξε για αυτή την απραξία, την αδράνεια στη Χαρτούμ, είναι κατάφορη εκεί βεβαίως η ευθύνη της Χαρτούμ, Ξέρουμε τις πολιτικές αποτυχίες και είναι πολλές αυτές. Τουλάχιστον να δανειστούμε ένα παράδειγμα για να δείξουμε σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια ήταν συνεχής και συνεπής. Έχει κάνει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαλύνει τα δεινά και τον πόνο του πληθυσμού στον Ταρφούρ. Το θέμα είναι εξύντλησε τα περιθώρια που είχε στη διάθεσή της. Ή δεν μπορούσε να είχε κάνει περισσότερο. Δεν ασκώ σε καμία περίπτωση κριτική προς τη Σουηδική Προεδρία. Όχι. Αλλά ανησυχώ και θέλω να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε τέτοιες περιστάσεις για να προλαμβάνουμε τα δεινά του κόσμου και ε, να μην υποφέρει. Λοιπόν, σας προτείνω να κάνετε αυτή την αποτίμηση. Ρίτα, μπορείτε να δεσμευτείτε αυτή τη στιγμή εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Ένωσης. Ε, Ευχαριστώ κύριε Γκέρενς. Σε μία πρόταση. Σήμερα συναντήθηκα με εκπροσώπους του Memorial των Ιγκούσων, της Ιγκουσετίας και μας είπε ότι από σήμερα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιληφθεί της κατάστασης. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ αργά, κατόπιν εορτής θα έρθουμε. Έχουν οξυνθεί πολύ τα πράγματα, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Κύριος Πρόντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μέρσελτ για την παρουσίασή της και την κυρία Αρνό. Είμαι νέος σε αυτή την υποεπιτροπή και ίσως να είμαι ακόμα και λίγο αφελής. Έχω όμως την εντύπωση ότι συχνά οι παρεμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παρεμβάσεις για τα συμπτώματα και δεν απευθύνονται στα αίτια, τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων. Γι' αυτό Κάποια ζητήματα πρέπει να επιληθούν μετά σε επίπεδο realpolitik. Νομίζω λοιπόν ότι μαζί με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και τα αίτια κάθε φορά. Έχω την εντύπωση ότι σε πολλές ε, περιπτώσεις ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση άσκησης εξουσίας που οφείλεται στην έλλειψη φυσικών πόρων και την αιμονή πολλών χωρών με την εξασφάλιση ακριβώς πρόσβασης σε φυσικούς πόρους. Αυτό οδηγεί στην ε, ανάδυση αυταρχικών ε, κυβερνήσεων, απολυταρχικών κυβερνήσεων. Αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημεία του κόσμου. Βλέπουμε μια διασύνδεση των απολυταρχικών κυβερνήσεων και την κατοχή φυσικών πόρων. Θα έπρεπε λοιπόν ίσως σε αυτό να σταθούμε και να κάνουμε και κάποιο είδους ανάλυση, μια μελέτη, να δούμε τι απαντήσεις μπορούμε να βρούμε συνολικά από το βήμα της δικαιοσύνης όχι να επικεντρωνόμαστε στις λεπτομέρειες, να δούμε σφαιρικά τα προβλήματα. Όχι μόνο να στεκόμαστε στο δράμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί είναι πολλά αυτά που μπορούν να λυθούν μέσω της διεθνούς δικαιοσύνης. Και όχι μόνο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά με οράματα ειρήνης κοινά και βεβαίως επιλύοντας προβλήματα ζωτικά όπως αυτό της πρόσβασης ε, στους φυσικούς πόρους, αυτό το πρόβλημα του Σουδάν, του Νταρφούρ. Νομίζω σε αυτή την προοπτική εντάσσεται και δεν είναι το μόνο. Θα πρέπει να απορρίπτουμε την επωνομαζόμενη τον, τον κινησμό μάλλον με τον οποίο Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα χωρών με εσωτερικές ε, διαταραχές. Και πολλές φορές το πρόσχημα είναι η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους. Να λοιπόν τι πρέπει να έχουμε κατά νου. Θα πρέπει να ασχολούμαστε με τη θεραπεία όχι μόνο των συμπτωμάτων, αλλά και των αιτίων της ε, κακής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κύριε Πρόντι. Πράγματι, οι φυσικοί πόροι και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζητήματα αλληλένδετα. Είναι σοβαρή η παρατηρήσή σα και θα πρέπει να το σκεφτούμε. Το τέλο τώρα του καταλόγου των αγορητών, δύο ακόμη συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Εάν συμφωνείτε, θα κλείσω εδώ τον κατάλογο των αγορητών. Γιατί έχουμε ακόμη δύο σημαντικά σημεία να δούμε. Την συζήτηση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και την σημαντικότατη μελέτη που έχει, οργανωθεί, που έχει ανατεθεί σε ένα Ινστιτούτο Μελετών. Κύριο Ντέβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ ε, την κυρία Σόλτ για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο σημαντική θέση καταλαμβάνουν ε, στις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας. Θα ήθελα να τη συγχαρώ, ήταν πραγματικά εξαίρετη. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια τα ερωτήματα. Αφού τα είπα όλα αυτά λοιπόν τώρα, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό αυτό έχουμε εμεί ω όπλο. Δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε ε, αυτοκίνητα, ούτε, ούτε ε, υποβρύχια, ούτε κανονιοφόρους, ούτε βομβαρδιστικά. Αυτό που έχουμε είναι η επιρροή μας. Είναι η γνώση που έχουμε και η ε, αυθεντία με την οποία μιλούμε και το κύρος ε, τα τεκτενόμενα στον κόσμο. Δηλαδή το τελευταίο που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς, το να το διανοηθούμε καν και το λέω επειδή τώρα ξεκινάει η Επιτροπή της Εργασίας, είναι να γελιοποιηθούμε στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, των Ηνωμένων Εθνών νομίζω απέτυχε διεθνώς. Και το γνωρίζουμε. Πραγματικά έχει γελιοποιηθεί. Είναι ε, περίγελος. Η δική μας Επιτροπή, από την άλλη, έχει εξαίρετα στελέχη με πάρα πολύ μεγάλη γνώση και θα πρέπει να κάνουμε τις παρουσιάσεις μας με τρόπο που να γίνεται πιστευτός και σεβαστός. Ό,τι και να λέμε θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας, μεγάλης γνώσης και κατανόησης του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων που εμείς ως κρατημέλη έχουμε αποφασίσει. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Θα πήρατε την επιστολή ε, που σας απίφθηνα για ένα θέμα στο οποίο δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω αλλά και στα πλαίσια της Σουηδικής Προεδρίας και της σημασίας που αποδίδει σε αυτά τα θέματα η Σουηδική Προεδρία. Δύο-τρία παράδειγμα. Ε, τα, δεν ξέρω αν τα έχετε υπόψη σας. Στο Μάλμο, στη Σουηδία, ή στην Ουψάλα, δεν θυμάμαι, στην Ουψάλα, συγγνώμη. Κάποιοι φοιτητές είπανε αν θεωρήσουν α πούμε ότι θέλουν να είναι εξάρτητοι. Δεν αναγνωρίζουμε τη Στοκχόλμη ω πρωτεύουσα και αρχίζουν και πυροβολούν δεξιά και αριστερά. Αντάτε. Είναι ε, πάντως αναγνωρισμένη χώρα η Σουηδία διεθνώ ε, και εμεί τι θα κάνουμε τώρα. Αν κάποιοι ξεσηκωθούν εκεί στην Ουψάλα ε, και θέλουν την εξαρτησία του, εμεί θα ανακατευθούμε. Φυσικά όχι. Αλλά καμιά φορά η Επιτροπή μα τίνει να το πράττει, στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν ήταν σε θέση να διακρίνει ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, όπου τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει συνθήκες και να γνωρίζουν ε, την εξαρτησία και την κυριαρχία των ανεξαρτήτων κρατών και επιμέρους ε, συμφέροντα τα κράτη-μέλη. Παράδειγμα, η Σρι Λάγκα. Η Σρι Λάγκα ήταν ενιαίο κράτος για 2.300 χρόνια, από το 400 π.Χ. μέχρι σήμερα. Ουδέποτε είχε υποστεί εισβολή ή ε, κατακαιρματισμό. Μπορεί να ήταν ε, απικία ε, και γνώρισε και Άγγλους και Πορτογάλους και Ολλανδούς, αλλά ως ενιαίο κράτος νήσος είναι μια λειτουργούσα δημοκρατία. Επίσης, 20 χρόνια πριν την κατάργηση της δουλείας, 15 από τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης ήταν απελεύθεροι ήδη η δούλη, η πάνω ε, από 100 χρόνια έχει εκλογές. Πρόσφατα μάλιστα έγιναν οι τελευταίες, και στο βορρά και στην Ανατολή. Τι προσπαθώ να σας πω τώρα, ότι ορισμένοι μπορεί να επικρίνουν τα κράτη-μέλη και την κατάσταση στη Σιλάνκα χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους ή να ξέρουν που πέφτει είτε τι ιστορία έχει η χώρα. Δεν μπορούμε ως Επιτροπή όμως να το πράττουμε αυτό και να θέλουμε να μας σέβεται και η διεθνή κοινότητα. Γιατί τα λέω και πάλι έτσι όλα αυτά, διότι η κατάσταση είναι τέτοια ε, που είναι, έχουμε 3, εκατομμύρια Ταμίλ που ζουν εκεί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και 2 εκατομμύρια είναι στο νότο, στις πόλεις. 1 εκατομμύριο στο βορρά. Εγώ μόλις γύρισα από το νότο και αν δείτε ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι και πιο εύποροι επιχειρηματίες είναι οι Ταμίλ. Το LTT έχει σκοτώσει περισσότερους Ταμίλ από ε, ε, Σιλανκέζους. Αυτά τα ξέρουμε όταν μιλάμε. Με ρωτάνε συνέχεια ο κόσμος από πού σας φέρανε σας τους ευρωβουλευτές. Και έρχομαι εδώ και να ε, σας υπερασπιστώ και εσάς και την Επιτροπή σας κυρία Πρόεδρε. Για αυτά που συμβαίνουν στη Σρι ε, από ορισμένα πράγματα που ξεστομίζει το κοινοβούλιο. Θα πρέπει να σταματήσουμε να τα κάνουμε. Κάνουν σωστά εδώ τα πράγματα, έτσι, για να μην μας θεωρούν ως... Πώς να το πω τώρα. Μια επιτροπή θερμοκέφαλων που λέει κάποια πράγματα τα οποία ε, μακροπρόθεσμα θα μετανιώσουμε γιατί θα είναι εις του Κοινοβουλίου. Γιατί και αυτά είναι τα μόνα μας όπλα επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεβά. Θυμήσατε ότι η επιτροπή μας χαίρει κάποιου κύρους και κάποιες αυθεντίες και θα πρέπει να το υπερασπιστούμε. Θα επανέλθουμε σε αυτή την κατάσταση της Ριλάνκα Λάγκα τέλη Σεπτεμβρίου. Έχουμε ακόμα ε, την κυρία Μπίλερ και μετά το Συμβούλιο. Ευχαριστώ την κυρία Αρνό. Ε, σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε, για την πρόσκληση στη Σοκχόλμη, για το άσυλο και τη μετανάστευση, για τη διάσκεψη. Σίγουρα θα το κάνουμε από ε, την ομάδα των Πρασίνων και την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Ερώτηση. Σε ποιο βαθμό εσείς η υπηρεσία σας συνεργάζεστε με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μια ακόμα ερώτηση. Πώς αξιολογείτε την πρόταση που λέει στην επόμενη Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει επίτροπος με αρμοδιότητα ανθρώπινα δικαιώματα, για να μην πω αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρόπου. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος για την ερώτησή σας. Πολύ καλή ερώτηση και πάρα πολύ συγκεκριμένη. Από πλευρά μου εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε περισσότερα και από το Ινστιτούτο της Βενετίας, από τη μελέτη που θα συζητήσουμε αργότερα. Η κυρία Κιόνκα έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ, εξ ονόματος Γραμματείας του Συμβουλίου. Πείτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε μετά από όλη αυτή τη συζήτηση. Α, η κυρία Χάμετσολτ, όχι, πρώτα η κυρία Κιόνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι εξίσου σύντομη με την προλαλή σας βουλευτή. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο ρόλο σας ως Πρόεδρε της Επιτροπής και στην υποπιτροπή αυτή τα καλύτερα για την περίοδο λειτουργία τη. Τρει σύντομε παρατηρήσει θέλω να κάνω για ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για. για τα σχόλια, προσθέτοντα μάλλον και εγώ τα δικά μου στα σχόλια τη Προεδρία και τη Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα για την υπογραφή και την κύρωση των διαφορών συμβάσεων Συμφωνώ απολύτως ότι η Επιτροπή ΚΟΧΟΜ και η πτυχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λειτουργούν ενθαρρυντικά για τα κάτι μέλη, να προχωρούν και ενεργά να κυρώνουν τις συμβάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι καθοριστικό για την αξιοπιστία μας στο διάλογο μας με τρίτες χώρες. Είναι κάτι που οι τρίτες χώρες συνεχώς ε, μας το ζητούν. Η δεύτερη παρατηρήσή μου έχει να κάνει με το Γκουαντάναμο και το κλείσιμο αυτού του στρατοπέδου. Είναι κάτι που ήδη ανέφερε η Προεδρία, να κάνω και εγώ δύο πλέον παρατηρήσεις. Η μία έχει να κάνει με το νομικό πλαίσιο και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο Γκουαντάναμο κάτι που παρακολουθούμε από το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συζητούμε και κλεισμένο των θυρών, έπειτα το 2006, λίγο αργότερα και στο πλαίσιο του διαλόγου με τους νομικούς μας συμβούλους και τους ε, εκπροσώπους του State Department, ξαναρχίσαμε να το συζητούμε και στα πλαίσια της προηγούμενης κυβέρνησης κυρίως, στη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αλλάξουμε λίγο την πορεία πλεύση αυτού του καραβιού, αν μπορώ να το πω έτσι. Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον Κουαντάναμο είναι ότι όταν εξελέγει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση και είχε την απόφαση για το κλείσιμο των ε, εγκαταστάσεων κράτησης στον Κουαντάναμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε θερμά την αποφασία αυτή της Αμερικανικής κυβέρνησης και Ουσιαστικά για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μα, όχι απλώ εγκρίναμε, αλλά προσφέραμε και τη βοήθειά μα. Ε, τα κάτι μέλη λοιπόν μετά από συζήτηση αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο θετικό περιβάλλον, υποστηρικτικό περιβάλλον ε, με κοινέ δηλώσει, αυτό που ανέφερε προηγουμένω και εκπρόσωπο τη Προεδρία για τον περασμένο Ιούνιο. Και κάτι που αποτελεί προσωπικό σχόλιο για τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνολικά αποφασίσαμε ω κράτη-μέλη να απευθύνουμε στι Ηνωμένε Πολιτείες την άποψή μα για το θέμα σε δύο πτυχέ. Πρώτα απ' όλα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα κάνουν τι απαραίτητε κινήσει στα πλαίσια ενό νόμιμου δικαστηρίου, κάτι που δεν νομίζουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί να. ένα ρόλο που μπορεί να αναλάβει αυτή η Επιτροπή. Και έπειτα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα λύσουν κάποια από τα προβλήματα που, των οποίων τα συμπτώματα αντιμετωπίζουν και τα ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Πρόντι. Προβλήματα λοιπόν που δημιουργήθηκαν από το σύστημα που δημιούργησαν οι ίδιες οι ΗΠΑ που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συμβάλει στην Task Force, την Task Force της διαδικασίας αναθεώρησης, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αν δεν χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του και να κλείσει τον Γκουαντάναμο, δεν θα έχουμε νίκη, αλλά μια πύριο, μια πύριο νίκη Αυτέ ήταν οι δύο μου και έχω και μια τρίτη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε του διαλόγου μα, τι διαβουλεύσει μα. Κάτι που επανειλημμένω αναφέρεται στην ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το συζητούμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Η αξιολόγηση για το διάλογο με την Κίνα που ανέφερε και η Προεδρία, η αξιολόγηση λοιπόν του διαλόγου αυτού είναι μια απόπειρα προ αυτή την κατεύθυνση. Εδώ αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι επικεντρωνόμαστε στον διάλογο με την Κίνα, αλλά Αφότου ξεκίνησε ο διάλογος αυτό πριν από 14 χρόνια, έχουν ξεκινήσει και άλλοι γύροι διαλόγων. Του ανέφερε προηγουμένω ε, σύντομα η Προεδρία. Εγώ, όταν ανέλαβα τη θέση αυτή πριν από δυόμιση χρόνια, υπήρχαν δύο ενεργοί διάλογοι και ένα παγωμένο τώρα. Έχουμε συνολικά 10, 12, 14, κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολο να κάνει κανεί τον σωστό λογαριασμό. Πάντω, εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι η αξιολόγηση τη Κίνα επικεντρώνεται μεν στην Κίνα, αλλά έχει στόχο να αποκομίσει διδάγματα και για τους νέους διαλόγους που έχουμε κινήσει. Οπότε προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό ως τρόπο βελτίωσης των ε, ενεξελίξεων διαλόγων και για το μέλλον μας. Είναι, αν θέλετε, μια, ένα πείραμα, μια δοκιμαστική διαδικασία για να γίνουν οι διάλογοι μας πιο αποτελεσματικοί. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. και Ευχαριστώ πολύ κυρία Κιόνκα. Η κυρία Άμερσολτ δέχτηκε πολλές παρατηρήσεις και ερωτήματα, αλλά και πολλά συγχαρητήρια προς τη Σουηδική Προεδρία για το πρόγραμμά της. Θέλετε το λόγο για να ολοκληρώσετε και πάλι, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω σε κάποια από τα κύρια ερωτήματα που ετέθησαν. Συνοπτικά. Πολλοί βουλευτές ρώτησαν ε, θέματα σχετικά με τη συνέχεια και τη συνέπεια ε, εθνικής πολιτικής και διεθνούς ρόλου και των δραστηριοτήτων μας σε διάφορα διεθνή φόρα. Ίσως να μου επιτρέπατε να πω τα εξή δύο. Πρώτον, θέλω να επαναλάβω ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης είναι και μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καθώς επίσης και σε άλλους μηχανισμούς που συνδέονται με συνθήκες, συμβάσεις και ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε διάλογο λοιπόν εκεί και αυξημένη ανταλλαγή εμπειριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε και τη διαφάνειά μας, ακριβώς την προβολή μας προς τα έξω για το τι κάνουμε, πώς σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και αυτό είναι ε, αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναθεώρηση της ε, ε, Συμφωνίας του Δουβλίνου. Επίσης, αναφέρθηκαν πολύ σε θέματα που έχουν να κάνουν με το mainstreaming που λέμε την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες πολιτικές της Ένωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη πρόκληση αυτό. Το αναγνωρίζουμε, αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να ε, το υλοποιήσουμε ενεργά στην πράξη και σε επίπεδο πολιτικής. Ε, μπορεί να συνδέεται αυτό με δύσκολες ε, επιλογές, έχουμε και διάφορα μέσα στη διάθεσή μας, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένοι τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Παράδειγμα, αυτό που είπε ο κύριος Χάουιτ για το πώς εργαζόμαστε στην Επιτροπή του Συμβουλίου, την COHOM, δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο αυτή η Επιτροπή με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, αλλά συνεργάζομαι με τους συναδέλφους που καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές στις επιτροπές τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την αξιολόγηση κατάστασης σε μια δεδομένη χώρα κάθε φορά. Επίσης θα έπρεπε να αναφέρω ότι συνεργαζόμαστε και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, παραδοσιακά στην Επιτροπή μας. Και στο Πολιτικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο κύριος Πρόντι μίλησε για την καταπολέμηση των αιτίων. Σίγουρα. Για να βελτιωθεί και η σχέση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναπτυξιακής πολιτικής. Με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να δούμε ε, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ε, της κάθε πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα άλλο τμήμα είναι να συνεργαστούμε για ε, τη δημιουργία δυνατοτήτων, έτσι, capacity building ονομάζεται αυτό η διεθνή δράση. Έγινε και μια συγκεκριμένη ερώτηση για τον Darfur. Θα μπορούσα να σας πω τώρα από πλευράς ευρωπαϊκής πολιτικής το εξής. Καταρχάς, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ταρφούρ μας απασχολεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μια πολύ στεναρή ε, θέση. Υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί που λειτουργούν και μπορούν να ψάξουν για ευθύνες για κατα... Ε, παραβιάσεων, ας πούμε, ε, καταπατήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το ένα μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι βεβαίως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν και την εντολή να εξετάζουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν ε, προκειμένου. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την εντολή, ας πούμε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ. Βεβαίως και θα συνεχίσουμε να θέτουμε αυτό το ζήτημα και άλλα ζητήματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικού δικαίου και λογοδοσίας σε περίπτωση παραβιάσεων των κανόνων αυτό. Κάτι άλλο που με ρώτησαν συγκεκριμένα για τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και πάλι είναι ένα ζήτημα αυτό όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ε, παγκόσμια. Πρώτα απ' όλα, πολύ ενεργά για να κυρωθεί το καθεστώς της Ρώμης. Σήμερα υπάρχουν πολλοί εταίροι που έχουν κυρώσει τη συνθήκη αυτή και προσβλέπουν στη συνεργασία με το δικαστήριο και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση το υποστηρίζει πάρα πολύ ως ανεξάρτητο δικαστήριο και φορέα. Ένα τελευταίο ίσως κυρία Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω όπως άρχισα. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνα, σας παραπέμπω στα όσα είπε τον Ιουλίο ο Πρωθυπουργός μου για τις μελλοντικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπουμε και εξετάζουμε μία σειρά θεσμικές ε, αλλαγές. Ε, και τελειώνοντας τα Σουηδικά, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά θερμότατα που μου επιτρέψατε να έρθω εδώ και να σας μιλήσω, να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας και επαναλαμβάνω ότι είμαστε απολύτως πρόθυμοι να συνεργαστούμε στο μέλλον με την Επιτροπή σας και με εσά προσωπικά για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε όλα αυτά που σήμερα σας παρουσιάσαμε και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που μας περιμένουν κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Ευχαριστώ κυρία Χάμερσχελτ. Είμαι ευτυχέστατος που μας διαθέσατε, ε, ευτυχέστατη που μας διαθέσατε τόσο χρόνο και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον παρίσταται η εκπρόσωπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Είμαστε ευτυχείς που σήμερα είσαστε τόσο πολύ άριθμοι στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ένα νέο θέμα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τακτικές συζητήσεις με το δίκτυο των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διότι είναι πολύ άριθμες οι σχετικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εκπροσωπούνται τώρα από τον Νικολά Ροζή της, ε, του Κλάπ της Ρώμης και και έχουμε και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συντονίζει τις εξωτερικές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον Νικολά Ροζή. Βέβαια, υπάρχει χώρος στο Προεδρείο και ευχαρίστως αν θέλετε ελάτε τουλάχιστον μπροστά. Ε, έχουμε διάφορα καθίσματα στις πρώτες σειρές τα οποία είναι στη διάθεσή σας. Okay. Thank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 θέλω να υποφεληθώ της ε, ευκαιρίας η οποία δίδεται και είναι πολύ σημαντική ε, για μας και ε, που μας επιτρέπει να διευρύνουμε τις σχέσεις μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της υποεπιτροπής και χάρηκα πολύ για τη συζήτηση με την κυρία Χάμερς Χελταρνό και Γιώκα που είναι θέματα σχετικά με αυτά που θα παρουσιάσω εγώ. Θα κάνω μία σύντομη εισαγωγή και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν για συνεργασία με αυτή την υποεπιτροπή. Καταρχήν όμως θέλω να σας πω ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Είμαστε μία ομάδα ε, περίπου 40 μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με τα θέματα της ε, προλήψεως και ε, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, βάσει της ε, ε, διεθνούς διακηρύξεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η οργάνωσή μας τονίζει την εξάρτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αλληλεπίδραση με τη δημοκρατία διότι προσπαθεί να προωθήσει ακριβώς ένα τέτοιο είδους δικαίου. Ποιοι, τι προσπαθεί προσπαθούμε να κάνουμε. And human rights at home and abroad as αλλά ε, ε, βασιζόμαστε στις αρχές που προαναφέρθηκαν από τους συναδέλφους και ε, πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πιέσει πολύ περισσότερο για να υπάρχει μη ένα σεβασμό των υποχρεώσεων που έχουν αναλυφθεί στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι θέματα που δεν μπορούμε να μετρήσουμε και πολλές φορές από διάφορους θεσμούς θεωρείται ως αυτοσκοπός και όχι ένας τρόπος για αλλαγή. Και οι μηχανισμοί για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν συνάδουν με την ε, προστασία των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, τρία θέματα που μας απασχολούν. Δηλαδή, καταρχήν να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, να υπάρχει μεγαλύτερο σοβασμός στις ανηλυμένες υποχρεώσεις για ανθρώπινα δικαιώματα και περισσότερη ε, διπλωματία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, πώς μπορούν αυτά να επιτευχθούν. Αυτό είναι το ερώτημα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθούνται σε όλους τους τομείς και είναι ένα βασικό θέμα της δραστηριότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν όμως ορισμένες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος που μπορούν να προωθήσουν το θέμα που μας απασχολεί. Καταρχήν, τη χρήση των οικονομικών μέτρων ε, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις και τις θεσμικές ε, αλλαγές για ε, την εισαγωγή μιας νέας συνθήκης. Πώς μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μία ανταλλαγή πληροφοριών ε, και να μπορεί να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στις διεργασίες αυτές ε, εφόσον ε, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπροσωπίες. Και τώρα θα δώσω το λόγο σε έναν συνάδελφό μου ο οποίος θα σας παρουσιάσει πιο συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, όλοι είναι σε ε, στενή συνεργασία με την υποεπιτροπή σας και άλλες επιτροπές και είχαμε μία θετική εμπειρία από τη συνεργασία αυτή και επίσης ε, ε, όσον αφορά τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και τι συνιστούμε να γίνει. Κατόπιν του, της διακηρύξεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα την οποία έχουμε ε, δημοσιεύσει και την οποία έχουν φαντάζομαι όλοι οι νέοι ευρωβουλευτές διότι υπάρχουν ε, ε, θετικές εξελίσεις στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται στο διάλογο εις τα ορισμένα τμήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, εις τα πλαίσια των περαιτέρω δράσεων. Επίσης όμως ε, η επιρροή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέτρων αυτών περιορίζονται λόγω ελλείψεως πολιτικής στηρίξεως ή έλλειψη ε, διοχετεύσεως στη σωστή οδό. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να εξασφαλιστεί ο σεβασμός για την προτεραιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων και εσωτερικά και εξωτερικά. Ο μεγάλος κίνδυνος βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι ε, απομονωμένα και οριζοντίως και καθέτος. Όσον αφορά την κάθετη πτυχή ε, είμαστε ε, απομονωμένοι αν δεν υπάρχει μια κοινή πιο ισχυρή θέση των κρατών μελών και όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής και οριζοντίως όταν δεν υπάρχει mainstreaming, δεν υπάρχει ενσωμάτωση και ε, δεν εντάσσονται εσωτερικά και εξωτερικά ή στην πολιτική, δηλαδή και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, στην πολιτική ε, μετανάστευση, στις συζητήσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Έχουμε δύο σημαντικές ε, συστάσεις που αναφέρονται στα θέματα αυτά της πολιτικής στηρίξεως και του mainstreaming Καταρχήν, το, η πρώτη μας σύσταση είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε την προσπάθεια διανοίξεως ενός πολιτικού χώρου για ε, συζητήσεις ε, μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών μελών, προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, διπλωματών τρίτων χωρών. Ε, και τονίζω ε, ότι είναι πολύ βασικό να συμμετάσχουν σε αυτά και ανεξάρτητοι προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρίτοι παρατηρητές για να υπάρχει μία συνεχής επαφή επιτόπου και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ε, μπορέσουμε να παρακολουθούμε καλύτερα την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αποφάσεων και των αποφάσεων των κρατών μελών. Ε, υπάρχει μια Αφρικανική Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει εκεί να υπάρχει μία ανεξάρτητη αξιολόγηση των ε, ε, ανεξαρτήτων αυτών θεσμών. Άρα τι πρέπει να προσπαθήσουμε θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων ε, της Προεδρίας, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ε, ανεξαρτήτων αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων και αυτό θα πρέπει να γίνεται πριν από τις διαβουλεύσεις ε, για πολιτική γυτνιάσεως και συζήτηση σε διάφορες επιτροπές και προτού οι αποφάσεις μπορέσουν να επηρεάσουν τις τρίτες χώρες, προτού ή κατά τις διαπραγματεύσεις ε, για εμπορικές ε, ε, συμβάσεις και για να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα τρόπο αναθεωρήσεως των μέτρων που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε επίσης να λάβουμε υπόψη τις διαβουλεύσεις οι οποίες πρέπει να οργανώνονται όποτε υπάρχει μία κρίση ή όποτε είναι αναγκαίο. Και αυτός ο διάλογος που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερομένους θα αυξήσει την πολιτική κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων σε όλες τις περιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο θα βελτιώσουν την ποιότητα των συζητήσεων αλλά επίσης θα καταστήσουν και τα κράτη πιο υπόλογα ε, και θα ε, βοηθήσουν τους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν και να υπάρχει μια καλύτερη αλληλεπίδραση με όλους τους ενδιαφερομένους.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 το δεύτερο σύνολο των συστάσεων αναφέρεται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, σε όλους τους τομείς ε, της κοινοτικής πολιτικής. Και το πρώτο θα είναι ε, να υπάρξουν μέλη σύνδεσμοι της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε αποστολές ε, προς τρίτες χώρες και σε διακοινοβουλευτικές ε, συνελεύσεις. Δηλαδή να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα είναι σύνδεσμος με τις άλλες επιτροπές και τις, ε, τους άλλους οργανισμούς. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινέ συνεδριάσεις με άλλες συνεδριάσεις, δηλαδή να υπάρχουν μεταξύ της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διαφόρων άλλων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοινέ συνεδριάσεις όπου θα αναφέρεται ε, το θέμα του, της διοχετεύσεως και οργανώσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει και μία κοινή επιτροπή μεταξύ της Επιτροπής Ελευθεριών και της Υποεπιτροπής ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ένταξή τους στις εξωτερικές πολιτικές. Για να τονίσουμε την ανάγκη που υπάρχει για να είναι υπόλοιγη και αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις τρίτες χώρες. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας ε, ε, ε, ε, διάλογος με τη Ρωσία παραδείγματος χάρη αν δεν ξέρουμε καν τι γίνεται στο επίπεδο που μας απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι να εστιαστούν συγκεκριμένες εκθέσεις εις ε, τα ανθρωπίνα δικαιώματα, στην καταπολέμηση τρομοκρατία, να υπάρχουν δηλαδή ε, διάφορα θέματα που άπτονται των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα οποία περιλαμβάνονται τις εκθέσεις αυτές και τέλος να υπάρχει μια γενική πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με την ε, συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής ε, ε, Δικαιοσύνης για να καθορίζονται τα ψηφίσματα, οι διακηρύξεις και οι δηλώσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μας δώσατε έπρεπε να είμαι πολύ σύντομος και πολύ γενικός γιατί εδώ εκπροσωπώ οι 38 διαφορετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αν θέλετε όμως τώρα θα έχουμε ε, τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ε, τριών οργανώσεων σε συγκεκριμένα θέματα και θα ξεκινήσουμε με τη Λίνα Νατούρα του Ευρωμεσογειακού Δικτύου που θα μας παρουσιάσει τα θέματά της. Ε, Ευχαριστώ. Το Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μέλος του γενικότερου δικτύου και απαρτίζεται από ε, οκτώ ε, οργανώσεις κρατών μελών της Μεσογείου ή κρατών που έχουν συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργασίας. Ξέρετε ότι το 1999 ξεκίνησε η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία και ε, ένας από τους διαλόγους ήταν διάλογος πολιτικής και ασφαλείας για να υπάρχει ένας κοινό χώρος ε, σταθερότητας και ασφάλειας ε, που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρασία. Το 1995 ξεκίνησαν αυτά, συγγνώμη. Το 2005 στη Βαρκελόνη, στη δεκάτη επέτειο, συμφώνησαν ε, τα συμβαλόμενα μέρη να προωθήσουν και την ισότητα των φύλων, να καταπολεμήσουν κάθε είδους διάκριση και να προωθήσουν ε, τη γυναικεία δικαιώματα. Ένα πενταετές πλάνο αποφασίστηκε. Και το 2006 στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, στην Υπουργική Διάσκεψη, ασχολήθηκε ακριβώς με την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών ε, στην κοινωνία και αποτέλεσε ορόσημο στα δικαιώματα των ε, γυναικών στην Ευρωμεσογειακή. 11 χρόνια μετά τη διακήρυξη της Βαρκελόνης υπήρξε ένας περιφερειακός μηχανισμός για την προώθηση ε, των γυναικείων δικαιωμάτων για πρώτη φορά και για την ισότητα των φύλων και συμφώνησαν εκεί και ε, όλοι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Αυτή η υπουργική διάσκεψη κατέληξη σε αυτό που ονομάζεται υπουργική απόφαση για την ενίσχυση ε, του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία. Το πλαίσιο της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι γνωστό σήμερα, το σχέδιο δράσης. Και πρόκειται να εφαρμοστεί από το 2010 στο 2006 στο 2010 με αιτήσιο μηχανισμό αναφοράς και τώρα έχει προγραμματιστεί επίσης η Υπουργική Διάσκεψη το ε, Νοέμβριο του 2012 στο Μαρόκο για να αναθεωρήσει να κάνει μια επισκόπηση των πεπραγμένων του προγράμματος δράσης. Δυστυχώς μέχρι το 2006 δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος στην Ευρωμεσογειακή ήταν μικρή συμμετοχή ε, των γυναικών και μικρές και προκλήσεις. Έλειπαν πολλές γυναικές ε, οργανώσεις και ακόμα και η Βαρκελόνη ασχολείται μόνο με τις γυναίκες στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας, χωρίς ειδική αναφορά, πούμε, στα δικαιώματα των γυναικών ε, και στις συμφωνίες σύνδεσης. Θεωρείται αυτό ένα πρόβλημα εσωτερικό της κάθε χώρας. Υπήρχε δηλαδή αυτή η τάση να θεωρούνται τα γυναικεία δικαιώματα ως ένα θέμα παραδοσιακό, ένα θέμα πολιτιστικό ή θρησκευτικό, οπότε και ε, εσωτερικό της κάθε χώρας. Και συνεπώς ε, δεν υπήρξε ούτε ενίσχυση των γυναικείων δικαιωμάτων ούτε mainstreaming στα διάφορα όργανα της Ευρωμεσογειακής. Το 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μια έκθεση για τα γυναικεία δικαιώματα και ε, ζήτησε ε, να γίνει και μια αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται όλα αυτά. Δυστυχώς δεν δόθηκε συνέχεια στις πρωτοβουλίες αυτές. Το πρόγραμμα δράσης σε διάφορα κράτη-μέλη περιλαμβάνει διμερή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ας και των ε, μεμονωμένων κρατών. Και βεβαίως ε, ο στόχος είναι να συμμετάσχουν όλοι στα προγράμματα δράσης, τα οποία δεν είναι νομικώς δεσμευτικά. Το περιεχόμενό τους και η υλοποίησή τους ε, εξαρτάται το επίπεδο δεσμεύσεων της, της επιμέρους χώρας. Με συγχωρείτε, πρέπει να σας διακόψω, γιατί όπως θα είδατε υπάρχουν πολλοί βουλευτές που φεύγουν. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε διάλογο, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, σύμφωνοι, τα ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των φίλων είναι σοβαρά, αλλά επειδή μας τελειώνει ο χρόνος, εάν θέλετε λοιπόν να έχουμε χρόνο και για διάλογο και συζήτηση, παρακαλούμε να συντομεύσετε. Ιδάλλως θα λείπουν οι συνάδελφοι και δεν θα υπάρξει καθόλου συζήτηση. Ίσως την επόμενη φορά να σας δώσουμε περισσότερο χρόνο για όλα αυτά τα ζητήματα και να διατηρήσουμε και την επαφή μεταξύ των διαφορετικών συναντήσεων. Απλώ, αλλά επειδή είχαμε προβλέψει έτσι κι αλλιώ δύο ομιλητέ, έχουμε πρόβλημα χρόνου. Θα έπρεπε να συντομεύσετε. Εντάξει, θα πω πολύ σύντομα αυτά που έχω να πω. Σύντομα, λοιπόν, μετά την Υπουργική Διάσκεψη του 2006, έχουμε και την Υπουργική Διάσκεψη του 2009, όπου θα υπάρξει αναθεώρηση του προγράμματος της ε, Ισταμπούλ. Μας απασχολεί ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου και της ε, Κοινοβουλευτικής ε, Συνέλευσης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το πώς μπορεί να οδηγήσει στην προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης διότι το έγγραφο τώρα ήταν αδύναμο και αυτό που θέλουμε είναι η στήριξη και η επιρροή του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να καταλήξουμε στην υπουργική διάσκεψη με ένα έγγραφο ε, ισχυρό και ένα πρόγραμμα δράσης που να έχει συγκεκριμένους σαφείς στόχους. Ε, επίσης και benchmarks, δείκτες δηλαδή, που να επιτρέψουν τη δημιουργία ενός ε, κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης. Υπάρχει και μια προσωρινή δήλωση που ετοιμάστηκε εν ώψη αυτή τη υπουργική διάσκεψη βάσει τη ανάλυση και τη μελέτη που κάναμε το 2006 με συγκεκριμένε συστάσει που μπορεί να σα βοηθήσουν να αποφασίσετε αν θα μα στηρίξετε ή όχι. Υπάρχουν αντίγραφα έξω από την αίθουσα των αντιγράφων. Θα ζητήσω από του αναπομείναντε ε, ομιλητέ να πάρουν το λόγο για δύο λεπτά καθένα. Ιδάλω δεν θα έχουμε καθόλου χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστούμε με Βερόνικα Σανταγκώσα που εκπροσωπώ το Human Rights Watch. Και πολύ σύντομα ήθελα να σχολιάσω τρει χώρε που αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωσία, Τουρκμενιστάν και Ουσμπεκιστάν. Για τη Ρωσία, καλωσορίζουμε τι έντονε αντιδράσει και του Ευρωκοινοβουλίου και τη Προεδρία του Συμβουλίου μετά την δραματική κλιμάκωση της βίας ε, και των βιοπριών στον ε, Βόρειο Κάφκασο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε εδώ όμω είναι ότι οι δολοφονίες αυτές δεν γίνονται στο κενό. Είναι σημαντικό να τις θέσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται της ε, έλλειψης δικαίου και της απτιμορρησίας για τις επίθεση κατά των ανθρώπ, της ανθρώπινης ζωής σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, η δέσμευσή μας με την ε, ρωσική κυβέρνηση να εργαστούμε κατά αυτής της ατιμορρησίας είναι σημαντική και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει, να πιέσει τη Ρωσία να αναλάβει σοβαρή δράση για να δώσει τέλος ε, στον κύκλο αυτό της βίας και των παραβιάσεων. Ένας συγκεκριμένο τρόπος που θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει εδώ είναι προωθώντας την πραγματική υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Τσετσενία. Υπάρχουν πάνω από 100 τώρα. Αν επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία πρέπει να υλοποιήσει τι αποφάσει αυτέ ε, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ήδη πέρυσι ε, επιμείναμε πολύ για τρεις από αυτές τις αποφάσεις και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο να επαναφέρει στο προσκήνιο μας στους διαλόγους με τη Ρωσία το ζήτημα αυτό. Θα ευχαριστούσαμε λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επιμείνουν για το ζήτημα αυτό. Για το Τουρκμενιστάν. πιο, το πιο πρόσφατο Συμβούλιο Γενικών και Εξωτερικών Υποθέσεων ε, επίσημα ενέκρινε μια συμφωνία, ενδιάμεσα συμφωνία με το Τουρκμενιστάν. Το Τουρκμενιστάν όμω είναι μια από τι πιο καταπιστικέ χώρε στον κόσμο. Και αυτό πραγματικά σοκάρει. Η γλώσσα για την ε, εμπορική αυτή συμφωνία δεν έκανε την παραμικρή μνήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά υπό το φω των ε, εντατικών συζητήσεων στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου συζητήσεων που μπλόκαραν επί σειρά ετών την σύναψη της συμφωνίας αυτής λόγω προβλημάτων με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο τον Απρίλιο και μετά τη συν τις εκπεφρασμένες δεσμεύσεις ε, του Επιτροπής και του Συμβουλίου προς το Ευρωκοινοβούλιο για τις σοβαρές ανησυχίες του Κοινοβουλίου για τον Τουρκμενιστάν και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί, μόνο τότε επιτράπει η συνάψη της συμφωνίας. Ιδίως για τους πολιτικούς κρατουμένους, τις περιορισμούς, τις μετακινήσεις και την απαγόρευση εισόδου των ειδικών ε, απεσταλμένων ε, του ΟΗΕ ή άλλων ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων της ε, Human Rights Watch, της ε, Διεθνούς Αμνηστίας και άλλων που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χώρα. Χρειάζεται εδώ λοιπόν διαμεσολάβηση προς την κυβέρνηση της χώρας <clears throat> και το Συμβούλιο καθώς και η Επιτροπή ανέλαβαν σαφείς δεσμεύσεις προς το Κοινοβούλιο να ασχοληθούν με τα προβλήματα αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζουμε λοιπόν θα επιτύχουμε πρόοδο σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει να δούμε και αποδείξει στα χέρια μα, για να πιστέψουμε ότι κάτι πετύχαμε. Και πάλι λοιπόν αυτό είναι ένα σημαντικό τομέα όπου ελπίζουμε το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα παραμείνουν πιστοί στις υποσχέσεις τους. Και η επόμενη σχέση συνεργασίας και εταιρική σχέσης που θα πρέπει να εξετάσει το Συμβούλιο του ερχόμενου μήνε είναι ακριβώ αυτό του Τουρκμενιστάν. Θα πρέπει λοιπόν το ζήτημα αυτό να παραμείνει ψηλά στι υποτεραιότητέ σα. Το Ουσμπεκιστάν τώρα είναι μια άλλη χώρα με ιδιαίτερα καταπιεστική κυβέρνηση, απολυταρχική, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει στενέ σχέσει. Είναι σημαντικό αυτό και γιατί λόγω του λόγω της διαδικασίας ε, που έχει προγραφεί για τον Οκτώβριο, θα δούμε τι θα γίνει με τις κυρώσεις που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή μετά τη σφαγή του 2005 και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εκπληρώθηκαν τα ανθρώπινα κριτήρια, τα κριτήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν τεθεί στον κυβέρνηση της χώρας, τα οποία για την ώρα μπορούμε εμείς να πούμε ότι δεν έγιναν σεβαστά. Όπως η απελευθέρωση πάνω από 12 πολιτικών κρατουμένων ε, για την πολιτική τους δράση, άτομα που εμποδίζουν την ε, κοινωνία των πολιτών στη χώρα να λειτουργήσει ομαλά. Επίσης, επαγορεύεται η είσοδος ε, των ειδικών απεσταλμένων του ΟΗΕ, αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα της Human Rights Watch, της Διεθνούς Αμνηστίας και άλλων. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο τα, τα κριτήρια αυτά ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, γίνονται σεβαστά και, κατά πόσο, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη μελέτη του αρχείου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χωρών αυτών. Να είμαστε αυστηροί. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο τελευταίο ομιλητή. Yeah. Yeah. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι λειτουργεί και το μικρόφωνο μου. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε και που δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω κι εγώ. Ε, έχω συντομεύσει ε, την παρέμβασή μου. Λάρς ε, δουλεύω για την CPN, την οργάνωση ε, για θέματα αναπηρίας και ε, ανάπτυξης και όπως καταλάβατε είναι μία από τις 38 οργανώσεις του ε, δικτύου και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στα θέματα της σύμβασης του ΙΕ για άτομα με αναπηρίες που ήδη έχει συζητηθεί στα πλαίσια ε, τη συζήτησή σας με τη Σουηδική Προεδρία, τουλάχιστον σε συντομία. Και η σύμβαση αυτή Τέθησε ισχύ ε, πέρυσι, την 1η Μαΐου και είναι συμβαλόμενα μέρος οι ευρωπαϊκές κοινότητες και αυτό είναι καινοτομία στο διεθνές δίκαιο. Όχι μόνο δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν προσχωρήσει που ε, παραδοσιακά υπογράφουν, κυρώνουν και εφαρμόζουν τη Συμβάση των Εθνών. Αυτή τη φορά έχουμε συμβαλόμενο μέρος εκτός από τα κράτη-μέλη και τις ευρωπαϊκές κοινότητες. Την Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε και το κοινοβούλιο σας και η Επιτροπή σας έχει να διαδραματίσει ρόλο στη διαδικασία κύρωσης, για να τη χαρακτηρίσω έτσι. Νομίζω νομικά ευσταθεί περισσότερο ο όρος ολοκλήρωση της σύμβασης. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν ολοκληρωθεί και ακούσαμε από τη Σουηδική Προεδρία ότι αναμένεται ακόμα κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας μέχρι τα τέλη του έτους Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε πλήρη διαδικασία ολοκλήρωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε την πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και το διάστημά της εφαρμογής και πώς θα μεταφραστεί στην πράξη αυτή η σύμβαση και όλες τις οι προοδευτικές ε, διατάξεις. Δυστυχώς δεν έχω την ευκαιρία να επεκταθώ, μάλλον χρειάζεται ξεχωριστή συνεδρίαση για να δούμε πώς θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες και στην Ευρώπη και αλλού. Δεν έχω όμως το χρόνο να αναφερθώ σε αυτό τώρα. Σύντομα θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε εσά και στην υποεπιτροπή σας να κοιτάξετε πολύ στενά τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θέλει και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ε, όσα συμφώνησε στη σύμβαση αυτή για τα άτομα με αναπηρία. Προς το παρόν αυτά και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία για εκτενέστερη συζήτηση του χρόνου ή ενδεχομένως και φέτος ακόμα αργότερα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος όλους τους ε, ομιλητές μας για αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ πολύτιμες ε, για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Μιλήσετε για το Ουσπεκιστάν, για τη Ρωσία. Αναφέρετε επίσης την υπουργική διάσκεψη και τα όσα μας αναμένουν το επόμενο διάστημα. Τι μας περιμένει. Επίσης τη Διεθνή Συμφωνία για τα άτομα με αναπηρίες. Όλα αυτά βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, τώρα ακολουθεί συζήτηση, δυστυχώς πάρα πολύ σύντομη, λίγων λεπτών, αλλά ε, αυτό που έχει εδώ σημασία ίσως είναι να δούμε ποια είναι η στρατηγική αξία αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Είπατε ότι χρειάζεται πολιτική υποστήριξη, mainstreaming κτλ. Τώρα καλό θα ήταν να περάσουμε στρατηγικές προτάσεις κάποια στιγμή για την υποεπιτροπή μας, γιατί είστε για μας στρατηγικοί εταίροι και ε, σύμμαχοι. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Και θα δούμε στη συνέχεια και σε επόμενες συνεδριάσεις πώς μπορούμε αυτή τη στρατηγική να την υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω ο τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν καταρτήσει μία διακήρυξη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που περιλαμβάνουν πολλά βασικά θέματα ε, και έχουν πολύ απαιτητικές ε, απαιτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λέγεται ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους. Ε, και δεν το πράττει. Συμφωνώ. Αλλά λέτε επίσης ότι για να εφαρμοστούν σωστά αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να διατηρηθεί η δύναμη των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις ε, το νέο κοινοβούλιο και θα χρειαζόταν ίσως μία διμερής απάντηση αλλά θα ήθελα να ξέρω τι εννοείται και ποια είναι η συγκεκριμένη σας σύσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουιτ. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι ο χρόνος δεν είναι μεν πολύ περιορισμένος και θα έπρεπε να θεωρήσετε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει το έργο της Επιτροπής σας. Σημείωσα τις κριτικές τις οποίες διατυπώσατε και πολύ θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας και στο μέλλον Θα ήθελα επίσης να σας πω πώς εργαζόμαστε σαν υποεπιτροπή και αν ε, θέλω να κατακρίνω τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις διαβάζοντας τη διακήρυξή τους και τις ε, δηλώσεις προς τις επερχόμενες προεδρίες ε, τα θέματα που θίγονται είναι αυτά τα οποία παρουσιάζονται εδώ και πέντε χρόνια. Αλλά καταρχήν όλοι συμφωνούμε με αυτά τα θέματα και το Κοινοβούλιο επίσης. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλα αυτά να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις στον κόσμο στον οποίο παλεύουμε και θα πρέπει οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να συνεργαστούν μαζί μας και με την Προεδρία για να καταρτήσουμε το πρόγραμμα του επομένου εξαμήνου και να το υλοποιήσουμε. Όσον αφορά ε, τους οικονομικούς πόρους τους οποίους αναφέρεται, ε, βεβαίως ε, είναι βασικά θέματα και δραστηριότητες όπου θέλουμε να συμμετάσχουμε και θα πρέπει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να μας ακολουθήσουν και όλοι να ακολουθήσουμε την ίδια οδό. Επίσης δεν ελέγχθη, αλλά στο παρελθόν, στο προηγούμενο κοινοβούριο, όταν το δίκτυο μας ε, το ζητούσε να έχουμε τακτικές συνεδριάσεις με το Προεδρείο της Υποεπιτροπής για να μπορούμε να συζητάμε σε μικρότερο κύκλο και ελπίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσετε και εσείς, γιατί απεδείχθη πολύ χρήσιμο ε, στη συνεργασία μας με την Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Εγώ προτείνω το εξής ε, σχετικά με τα, τη χρήση των επομένων 45 λεπτών. Να ακούσουμε μία εισαγωγή σχετικά με τη μελέτη είναι το ίδιο θέμα το οποίο παρουσίασε ο κύριος Τιερή, το mainstreaming δηλαδή. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 7. διότι η Υποεπιτροπή έχει αναθέσει μία μελέτη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενσωμάτωσή τους στις εξωτερικές σχέσεις και ο καθηγητής Φλωρόνς Μπενουά Ρούμερ, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της IUC στην Βενετία και που στο παρελθόν ήταν επικεφαλής του Πανεπιστημίου Ρομπέρ Σουμάν στη, στο Στρασβούργο και ο, ο, ο καθηγητής Χόρστ Φίσερ που είναι πρόεδρος του IUC θα μας παρουσιάσουν το θέμα αυτό. Και οι δύο κύριοι αυτοί είναι εδώ και εκπροσωπούν ε, τους οργανισμούς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαστε σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη που ετοιμάστηκε από το ΛΙΟΚ, όπως ονομάζεται, το Διαπανεπιστημιακό Ευρωπαϊκό Κέντρο για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκδημοκρατισμού. Η έδρα βρίσκεται στη Βενετία και εκεί συνεργάζονται 41 πανεπιστήμια ε, με σκοπό να προωθήσουν την εκπαίδευση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πραγματοποιήσουν μια σειρά μελετών και ε, αναλύσεων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι πήραμε την ε, μας αποδόθηκε η μελέτη αυτή μετά το διαγωνισμό του Ευρωκοινοβουλίου για το ζήτημα των mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εμείς λοιπόν αναλάβαμε τη μελέτη αυτή βάσει του διαβολισμού, της διαδικασία που οργανώθηκε. Στις 4 Μαΐου 2009 ολοκληρώθηκε η μελέτη, μελέτη που πραγματοποιήθηκε από δεκάδες ε, εκπαιδευτές, ε, καθηγητές, μελετητέ του κέντρου μα ένα έγγραφο που ετοιμάστηκε με σκοπό να αξιοποιηθεί από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή και διεξάχθη μετά από πολλέ συνεντεύξει με υπαλλήλου, στελέχη του Κοινοβουλίου, τη Επιτροπή, του Συμβουλίου και με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ε, και εδώ θα εκπροσωπήσω του συναδέλφου μου για να ανακεφαλώσω το περιεχόμενο τη μελέτη αυτή. Ήθελα να επιμείνω κυρίω στις συστάσει που θα μπορούσαμε να απευθύνουμε προ το Ευρωκοινοβούλιο για να βελτιώσει ενδεχομένω το mainstreaming στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι εξωτερικέ του σχέσει. Το πρώτο ερώτημα που θέσαμε στου εαυτούς μα είναι τι ε, σημαίνει ακριβώ ο όρος mainstreaming. Για μια Γαλλίδα είναι ένα όρος ιδιαίτερα περίπλοκος γιατί δεν υπάρχει ακριβή μετάφραση του όρου στα γαλλικά. Μπορεί να μιλήσει κανείς για διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν είναι ακριβώ το ίδιο το νόημα. Νομίζω όταν μιλάει κανεί για mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ουσιαστικά εννοεί το εξή. Ε, ε, να ε, επικεντρώσει τη συζήτηση που γίνεται στην κοινωνία γενικώ για διάφορα ζητήματα τα ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώ, το κέντρο αυτό ενδιαφέροντο. Δηλαδή από το περιθώριο να περάσει στο κέντρο ενδιαφέροντο τη κοινωνία ε, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διεθνώ, ο όρο του mainstreaming στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημαίνει για τους διεθνείς οργανισμούς, μια στρατηγική που σκοπό έχει να ενσωματώσει με θελημένη προσέγγιση την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο των δραστηριοτήτων, στο σύνολο των πολιτικών ενεργειών. Ο στόχος λοιπόν του mainstreaming επιτυγχάνεται όταν ο διεθνής οργανισμός δεν αρκείται πλέον να ασχολείται με την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένε ε, δραστηριότητες και προσπάθειες, αλλά όταν η μεθοδολογία του πρότυπου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων του οργανισμού, του εν λόγω οργανισμού. Όταν η μεθοδολογία, δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικά εμποτίζει την ε, ε, νοοτροπία ολόκληρη, τη φιλοσοφία του διεθνούς οργανισμού. Ε, με τη γέννηση του όρου αυτού, εφόσον τη μελετήσαμε, είδαμε ότι ξεκίνησε η χρήση του όρου στον ΟΗΕ, όπου υποστηρίχθηκε ιδιαίτερος από το Γενικό Γραμματέα Κόφι το 1989, όταν ο κύριος το 1999 όταν ο κύριος Ανάν ε, μίλησε για την ε, ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του ΟΗΕ. Η UNICEF ήταν ο πρώτος, το πρώτο δικαιωμένο σώμα του ΟΗΕ που χρησιμοποίησε ευρέω τον όρο αυτό. Δεν θα επανέλθω σε αυτό. Εάν θέλετε λεπτομέρειε περισσότερε μετά, μπορείτε να τις ζητήσετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση ε, ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση από τη δεκαετία του 2000. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε ακριβώς στην πολιτική του και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια από ό,τι για τον ΟΗΕ, διότι η διατήρηση της ειρήνης είναι από τις κατεξοχήν ε, αποστολέ του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά ήταν ένα οικονομικό οργανισμό που σκοπό είχε να βελτιώσει την ευημερία, την οικονομική ευημερία των πολιτών τη Ευρώπη και να ευνοήσει τη δημιουργία οικονομικής ελεύθερης αγοράς. Δεν είναι ακριβώς ίδιος ο σκοπός των διοργανισμών. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει mainstreaming σε πολλές από τις πολιτικές της. Ε, ε, στην πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εμπορικών πολιτικών, των μεταφορών της ενέργειας και το καθεξής. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δέσμευση για το mainstreaming στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι σημαίνει. Σημαίνει ακριβώς ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συστηματικά θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των πολιτικών της Ένωσης. Είτε αφορούν τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε διαφορετικού τομεί όπω εξωτερικέ σχέσει ή εξωτερική διάσταση όλων των πολιτικών, των εσωτερικών, όπω το άσυλο και η μετανάστευση, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικέ υποθέσει, η ενέργεια και ούτω καθεξής. Προφανώς το Ευρωκοινοβούλιο είναι μια από τις κινητήριες δυνάμεις της πολιτικής αυτής του mainstreaming ε, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το 2007 στη δήλωση για τα, ανθρώπινα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιμένει στην ανάγκη να περάσουμε σε mainstreaming στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων το Κοινοβούλιο. Επίση, στην ετήσια, ετήσια έκθεση του του 2007 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω, επιμένει το Κοινοβούλιο στην ανάγκη ενίσχυση τη ΠΕΣΚ, και τη εξωτερική πολιτική ασφάλεια και άμυνα, η οποία συχνά δυσχεραίνεται από τι εγωιστικέ ε, τάσει των ε, κρατών μελών και ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προτεραιότητα. Και για να προωθήσουμε την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω στόχο τη ΠΕΣΚ, θα πρέπει αυστηρός να επιμένουμε στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών. Ο ρόλος λοιπόν του Κοινοβουλίου ανέκαθεν ήταν να στηρίζει την πολιτική του mainstreaming και να εξακριβώνει ότι η πολιτική αυτή ακριβώς υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η διάγνωσή μας, θα είμαι αρκετά σύντομη, όπως είδαμε από την αρχή της απογευματινής αυτής συζήτησης, η πολιτική του mainstreaming ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εξωτερικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπαρκτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όργανα και εργαλεία για να υλοποιήσει την πολιτική αυτή του mainstreaming και διαθέτει επίσης συγκεκριμένα μέσα. Το mainstreaming λοιπόν και η πολιτική του υπάρχουν, υπάρχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της. Υπάρχει από το 2001 λοιπόν ένας αριθμός εγγράφων, σημαντικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων, εκθέσεων, συμπερασμάτων, τα οποία έχουν ετοιμαστεί από τα διάφορα θεσμικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όλα αυτά τα μέσα ορίζουν το νόημα του mainstreaming. Τα έγγραφα αυτά αρχικά αφορούσαν κυρίως τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή την ΠΕΣΚ, την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, και επιτάω έχω ήταν να η πολιτική αυτή και να έχουμε μια διευρυμένη προσέγγιση σε όλες τις πολιτικές, όπως την εξωτερική διάσταση του πρώτου και του τρίτου πυλώνα. Η εξωτερική διάσταση του πρώτου και του τρίτου πυλώνα μπορεί να αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τη συνεργασία ε, στα ποινικά ζητήματα, το άσυλο και τη μετανάστευση και το καθεξής. Τα μέσα που η Ένωση διαθέτει για να κάνει mainstreaming ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ποικίλα. Τα έχουμε σχολιάσει ξανά και ξανά, κάποια είναι πιο γενικά, κάποια πιο ειδικά. Υπάρχει ο διάλογος που είναι ιδιαίτερα προσφυλή στα τρίτα κράτη, σχεδόν όλα τα τρίτα κράτη. Υπάρχει ένας αριθμός κατευθυντήριων γραμμών που ετοιμάστηκαν προκειμένου να δοθούν κατευθύνσεις στις σχέσεις με τα τρίτα κράτη, όπως ε, τα βασανιστήρια, η απαγόρευση των βασανιστήριων, η απαγόρευση της θανατικής ποινής, η υπεράσπιση των, ε, των ατόμων που δρούν ως ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και υπάρχουν ρήτρε στι εμπορικέ συμφωνίε που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τι συμφωνίε αυτέ ή να αναλάβει κυρώσει, να επιβάλλει μάλλον κυρώσει, σε περίπτωση που τα συμβαλόμενα κράτη δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν επίση οι συμφωνίε των γενικών προτιμήσεων και υπάρχει και το περιβόητο αυτό μέσο τη Ευρώπη για τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οικονομικό εργαλείο, αλλά επιτρέπει να υλοποιηθούν οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση στην σημασία του mainstreaming. Νομίζω ότι τα εργαλεία λοιπόν υπάρχουν από θεσμική άποψη στα θεσμικά όργανα. Επίση υπάρχουν, ξέρουμε ότι το Συμβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο για την πρόθεση του mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χάρη στον Γενικό Γραμματέα του και τον ε, προσωπικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, τον είπα το εκπρόσωπο. Δεν θα επιμείνω και στον ουσιαστικό ρόλο του Γενικής Γραμματείας, του προσωπικού. Αυτά είναι γνωστά σε επίπεδο του Συμβουλίου, είναι όμως πολύ σημαντικά για την διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τον συντονισμό των δράσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες πολιτικές και στην εξωτερική τους διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή και εκείνη εμπλέκεται σοβαρά στην όλη διαδικασία ε, λόγω της συνεργασίας που έχει εγκαθιδρυθεί με την ΔΕΣΚ, με το Συμβούλιο ε, και τον κοινό καθορισμό πολιτικών από πλευράς του, ιδίως των περιφερειακών πολιτικών. Επιτροπή έχει ως βασική της αποστολή να υπενθυμίζει και το κάνει την σημασία του mainstreaming στα διάφορα στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο και αυτό ε, συμβάλλει στην πολιτική του mainstreaming, λόγω χάρη μέσω της συμμετοχής τους της αποστολές της ε, παρακολούθησης εκλογών ή με ψηφίσματα που διαρκώς υπενθυμίζουν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με εκθέσεις που ετοιμάζονται, ιδίως την ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάστασή τους. Ξέρουμε πόσο η δράση του Κοινοβούλιο εδώ είναι σημαντική, διότι το Κοινοβούλιο είναι ο δρόμος της Ευρώπης, είναι ακριβώς η νομιμοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της. Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά αυτά που μας είπαν ε, όσοι ερωτήσαμε. Και στη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας συνεντεύξεων ε, έχουμε μια παρατήρηση που συχνά επανέρχεται. Η έλλειψη συνοχής μεταξύ τη εσωτερική και εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ε, κρατών μελών ξεχωριστά. Κάτι που αποδυναμώνει την ε, τοποθέτηση πολλέ φορέ σε, σε πολλέ περιπτώσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ζητήματα διεθνή, όπω αυτά που έχουν να κάνουν με το Διεθνέ Δικαστήριο. Ή η ανάγκη ενίσχυση του γεωγραφικού και του θεματικού σκέλου ή του πολυμερούς και του διμερούς. Πρέπει λοιπόν στη λειτουργία του mainstreaming να ενισχύσουμε κι άλλο, κι άλλο την συνοχή, τον παράγοντα της συνοχής σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό για τον επιπλέον λόγο ε, που αντιλαμβανόμαστε ότι η υλοποίηση των πολιτικών του mainstreaming χρειάζεται να, απαιτεί να είμαστε συστηματικοί και να δίνουμε διαρκή προσοχή στην ε, εξέλιξη της διαδικασίας. Η διαδικασία θα πρέπει λοιπόν να είναι συστηματική ε, για όλα τα σκέλη. Επίσης, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ατόμων που ακούσαμε σε συνέντευξη, τα πολιτικά δικαιώματα και κοινωνικά δικαιώματα λαμβάνονται υπόψη, αλλά όχι τα οικονομικά και πολιτιστικά αναγκαστικά. Επαναλαμβάνω τα λόγια των ανθρώπων που μας μίλησαν για τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αυτό το πλαίσιο πολλές ήταν με κυβερνητικές ε, οργανώσεις που εξέφρασαν την επιθυμία να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Επίσης, πολλοί μας είπαν ότι μπορεί να υπάρξει περισσότερη, καλύτερη υλοποίηση μάλλον του mainstreaming στην εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιούνται με ακόμη πιο συνεκτικό τρόπο και πιο συντονισμένο τα οικονομικά, τα περιβόητα οικονομικά εργαλεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδίω και τον εκδημοκρατισμό. Για να ολοκληρώσω με τη διάγνωση που κάναμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πολιτική mainstreaming για τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως κρίμα είναι που δεν ε, έχει δώσει συστηματική έμφαση στα μέσα αυτά που εκδιπλώνει, στα συγκεκριμένα εργαλεία και ιδίως κατά την υλοποίηση των πολιτικών. Τώρα, υπό το φως των όσων ακούσαμε, Στι συνεντεύξει, θελήσαμε με κάθε ταπεινοφροσύνη να διατυπώσουμε έναν αριθμό συστάσεων, συστάσεων προς το Κοινοβούλιο, συστάσεων που μας προτάθηκαν ακριβώ από τα άτομα με τα οποία συζητήσαμε. Και δώσαμε κι εμείς τη συγκατάθεσή μας ε, στις προτάσεις τους. Σε θεσμικό επίπεδο πρώτα απ' όλα. Κάποια άτομα, το μεγαλύτερο μέρος των ε, ανθρώπων με τους οποίους συζητήσαμε εκτιμούν ότι σήμερα χρειάζεται μια κεντρική δομή που να διασφαλίζει την συνοχή της πολιτικής mainstreaming στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κεντρική δομή που να ετοιμάζει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις προς τα υφολοθεσμικά όργανα, προκειμένου να βελτιώσουν την πολιτική του mainstreaming. Κάποιοι θεώρησαν αναγκαίο να δημιουργηθεί εν μια θέση ε, Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου αυτού θα περιλάμβανε τη διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην εξωτερική διάσταση όλων των εσωτερικών πολιτικών. Επίσης θα αναλάμβανε αυτός ο Επίτροπος τον συντονισμό με τον εκπρόσωπο της ε, ΚΕΠΑ και με τους ε, υπόλοιπους επιτρόπους σε ό,τι αφορά τον ε, τομέα αρμοδιότητάς τους. Έπειτα αυτός ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ήταν μεταξύ των υπολείπων υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό του σε εσωτερικό επίπεδο, ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ εσωτερική και εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα, αλλά φάνηκε κάπως ουτοπική σε κάποιους άλλους. Υπήρξαν αντιδράσεις θετικότατες ε, προς την πρόταση αυτή, αλλά και αρνητικότατες. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι πρόκειται για μια ιδέα μάλλον ουτοπική. Διότι μιλάμε για επικάλυψη των όσων ήδη υπάρχουν σε επίπεδο Συμβουλίου και Επιτροπή, αλλά και ενό άλλου θεσμικού οργάνου, το Επιτρόπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Πάντως αυτή η ιδέα του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μα άρεσε πολύ. Άλλα μέτρα, λίγο πιο ρεαλιστικά, θα μπορούσαν να ληφθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία για να διευκολυνθεί το mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε την ενότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γενική Διεθνή Ρέλεξ. Υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες εκεί, οι οποίες είναι διασπαρμένες από υπηρεσία σε υπηρεσία. Σας μίλησα για την ιδέα του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά αν θέλουμε η υπηρεσία αυτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ασκεί τι εξουσίε τη στην εσωτερική εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, προσωπικού. Επίσης θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την αναβάθμιση της υπηρεσίας σε διεύθυνση ενδεχομένως ε, αυτοκέφαλη, η οποία να μπορεί να βελτιώσει την προβολή τη υπηρεσίες των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την όλη πολιτική, την βούληση αυτή να γίνει mainstreaming στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλο προτινόμενο μέτρο σε κάθε γενική διεύθυνση πιστεύουμε και η πρόταση αυτή μας έγινε επανειλημμένος. Θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν σε κάθε γενική διεύθυνση της Επιτροπής μία υπηρεσία η οποία να ασχολείται ακριβώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι εξειδικευμένα υπεύθυνη για το mainstreaming στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ασχολείται με τα σχετικά ζητήματα, τις σχετικές υποθέσεις. Να οργανώνει το mainstreaming στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εν λόγω Γενικής αλλά και στις διάφορες δραστηριότητες των διαφόρων γενικών διευθύνσεων μεταξύ τους. πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που αφορούν την εκχώρη, τις αντιπροσωπείες, τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, επικεφαλής των αντιπροσωπιών που διδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι αντιπροσωπείες αυτές θα έπρεπε ακόμη περισσότερο και από στρατηγική άποψη να συμβάλλουν στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να οργανώνονται λοιπόν συναντήσεις συντονισμού με τους διαφόρους επικεφαλής αντιπροσωπιών των κατών μελών, προκειμένου καλύτερα και περισσότερο να ληφθούν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλιστεί το mainstreaming άλλα μέτρα. Εκφράστηκε η επιθυμία, η περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων για τις ε, θέσεις κλειδιά στην Επιτροπή να περιλαμβάνουν και κάποιε ειδικέ γνώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή κάποιο γενικό διευθυντή ή κεφαλή υπηρεσία να μην μπορεί να προσληφθεί αν δεν έχει κάποιε ελάχιστε γνώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν και άλλα μέτρα, μέτρα εκπαίδευση εδώ που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με αυτό που προαναφέρθηκε. Μπορούν πολλά να διδαχθούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο προσωπικό που εργάζεται επί τόπου. Νομίζουμε λοιπόν ότι μπορεί να καταρτιστούν καλύτερα στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα άτομα αυτά που ασχολούνται με τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδού για την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα στο Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος του προσωπικού προσώπου του Γενικού Γραμματέα του προσώπου. Ε, μας φαίνεται καθοριστική σημασία σε αυτό γιατί η δράση του προσωπικού προσώπου στον χώρο της ΚΕΠΑ είναι καθοριστικός, παίζει ρόλο ζωτικό για το mainstreaming και τη διάδοση της ε, όλης κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ρόλος λοιπόν αυτός πρέπει να ενισχυθεί, να ενισχυθεί το στάτους του συγκεκριμένου ατόμου, το πολιτικό του βάρος, ώστε να διασφαλίσουμε το mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποκτήσει την απαιτούμενη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδού οι θεσμικές μου λοιπόν συστάσεις. Οι συστάσεις τώρα για τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η εξή. Νομίζω πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος, διάλογος που όπως είπα είναι ούτως ή άλλως προσφυλής στα τρίτα κράτη, πάνω από 30 διάλογοι βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το είπε και η κυρία Αρνό προηγουμένω. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουν οι διαδικασίε αυτέ διαλόγου και αν ε, μιλήσει κανεί με όσου συμμετείχαν στους διαλόγους αυτούς, ε, ακούει ότι υπάρχει κάποια απογοήτευση για την ανεπάρκεια, όχι απουσία, αλλά ανεπάρκεια στην οργάνωση των διαλόγων αυτών. Θα ήθελαν οι διάλογοι αυτοί να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα, ώστε να γίνονται συζητήσει όχι επιφανειακέ, αλλά συζητήσει ει βάθο. Να περιοριστεί ο αριθμό των θεμάτων για να ενισχυθεί ακριβώ ε, αντιστρόφως η ουσία των συζητήσεων. Και επίση να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφορών τρεχών των διαλόγων. Αυτά για τους διαλόγους, ε, για τις κατευθυντήριες γραμμές όλοι βεβαίως τις εκτιμούν τις θέλουν, όμως πρέπει και αυτές να ενισχυθούν. Ιδίω η χρήση τους. Η χρήση τους πρέπει να αξιολογείται. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία, να αξιολογούνται σε τακτά χρονοκαδιαστήματα οι κατευθυντήριες γραμμές, τα guidelines και οι αξιολογήσεις αυτές να αξιοποιούνται με τη σειρά τους για να καθορίζονται τα ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν στους επακόλουθους διαλόγους ώστε να, γι, να δίδεται έμφαση στα σημεία κλειδιά, τα καθοριστικά σημεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι αξιολογήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και για την καλύτερη επιλογή των ε, προγραμμάτων που θα επιλεγούν από το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό. Οι κατευθυντήριες γραμμές επίσης θα πρέπει να καλύπτουν και τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, ώστε ε, η αρχή του αδιέρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχώ αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβάλλονται από το Ευρωκοινοβούλιο, που είναι από του βασικού υπερασπιστέ του αδιέρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά να μπορέσουν χειροπιαστά να υλοποιηθούν στι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να πω ακόμη κάτι και για το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την Τρόπινα ε, Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό εργαλείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του mainstreaming του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στου διάφορου τομεί δραστηριότητα που χρηματοδοτούνται, ιδίω στη χρήση των κατευθυντήρων γραμμών και του διαλόγου προκειμένου να καθοριστούν τα προβληματικά σημεία για τη χρηματοδότηση δράσεων. που προσανατολίζονται να βελτιώσουν την κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ οι λίγες συστάσεις που θέλαμε να σα ε, εκφράσουμε τώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του ιδρύματό μα για να προσθέσει ενδεχομένω ορισμένα πράγματα σε αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και είναι κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε αυτή τη μελέτη. Δύο σημαντικά θέματα συμβαίνουν. Η συνθήκη της Λισαβόνας ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστεί πράγμα το οποίο θα είναι μια ευκαιρία για την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σκεφτούν πώς θα οργανώσουν την εργασία τους στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετά η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ίσως έναν νέο επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τα θα ακούσουμε μια τέτοια συζήτηση. Ο Δόκτωρ Φίρισερ, Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να είμαι σύντομος διότι έγινε μία σωστή συνόψιση της μελέτης. Πρέπει όμως να σας πω ότι στην ομάδα η οποία κατάρτισε την μελέτη ασχοληθήκαμε με το θέμα της τεχνολογίας σχετικά με το mainstreaming. Υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά την Ευρώπη στο θέμα αυτό ε, και πρέπει να δούμε τι σημαίνει το mainstreaming και με τι μεθοδολογία εφαρμόζεται για να δούμε πώς δράει η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Συζητήσαμε επίσης και αυτό είναι το επιστέγασμα της ε, συστάσεως να γίνει ένα, ε, μια εξέταση, ένα screening του mainstreaming ασχέτως αν μπορέσει αυτό να γίνει ολοκληρωτικά αλλά μια, ένα τέτοιο screening πρέπει να γίνει σχετικά με το mainstreaming και τέλος το θέμα το οποίο ε, σχολιάστε τελευταία δηλαδή τον Επίτροπο για για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεδομένη ε, της οικονομικής κρίσεως και των κλιματολογικών αλλαγών και εφόσον αυτά τα δύο θέματα δεν μπορούν να απαντηθούν ικανοποιητικά χωρίς ε, την εμπλοκή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν μέχρι στιγμή στο mainstreaming ακόμη και για το περιβάλλον. Υπάρχουν ορισμένα πρόσφατα ε, έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα εξετάζονται λιγάκι στο ποδάρι και θα πρέπει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εμπλεκόμενα πανεπιστήμια να μπορέσουν να αποδείξουν ότι οι δύο αυτοί βασικοί τομείς, η οικονομική κρίση και η κλιματολογική αλλαγή πρέπει να συμπαρασύρουν συζήτηση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη σημαντική παρατήρηση. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, Νομίζω ότι το mainstreaming ε, σχετικά με την ισότητα των ε, φύλων αποτελεί ε, ένα παράδειγμα. Δεν υπήρξε πάντοτε επιτυχής αυτή η προσπάθεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ έχουμε δεσμευτεί για την ισότητα των φύλων και για το mainstreaming των φύλων. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσω την την ε, ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει. Θα ήθελα να ξέρω τι έχει να πει ε, ο κύριος Τιερή, αλλά δεν θα του διαθέσουμε τόσο χρόνο στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, καθότι η κυρία Αρνό προηγείται. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι υποθέτω ότι αυτή η μελέτη θα οδηγήσει σε πιο εμπεριστατωμένες μελέτες. Είναι πολύ ενδελεχής, πολύ σαφής και δίνει μία πολύ καλή παρουσίαση των εξελίξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να τονίσω μερικά βασικά θέματα συγκεκριμένα που μας απασχολούν και που είναι υλοποιήσιμα. Οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις έχουν γίνει από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι όλοι οι αρχηγοί αποστολών τώρα έχουν ε, καθορίσει έναν υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει και ένας πολιτικά υπεύθυνος και ένας τεχνικά υπεύθυνος διότι πιστεύαμε ότι θα περιοριστούμε στο θέμα της συνεργασίας αλλά τώρα θέλουμε να τονίσουμε και τον πολιτικό διάλογο και γι' αυτό υποκινούμε τις αντι να ε, συσφίξουν τη σχέση μεταξύ πολιτικής ε, και τεχνικής πτυχής, να έχουμε συνεργασίες και συναντήσεις με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με τα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο γίνεται τώρα συστηματικά ε, πριν οργανώσουμε συζητήσεις με τρίτες χώρες. Μία πολύ βασική ιδέα, αλλά αντίθετα με αυτά τα οποία είπε η κυρία Φλωρόρο είναι εάν οι τρίτες χώρες ενδιαφέρονται να έχουν συζητήσεις μαζί μας διότι εμείς θέλουμε να συζητάμε μαζί τους, αυτοί όμως όχι τόσο. Δηλαδή δεν έχουμε απέναντί μας τους ε, συνομιλητές τους οποίους επιθυμούμε. Υπάρχει ένα φράγμα του Υπουργείου Εξωτερικών και υπάρχει η γραμμή του κόμματος, η party line, ενώ θα πρέπει να έχουμε τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων ε, Εσωτερικών ε, Δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε και τέλος Όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, είναι κάτι όπου θεωρητικά είπαμε ότι πρέπει να ισοσχελίσουμε τα πράγματα γιατί πολλά έχουν γίνει ε, όσον αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, αλλά εφόσον είμαστε οι πρώτοι δωρητές ε, ταξί των κρατών της Ευρώπης και από την άλλη μεριά λέμε ότι δεν προχωρούμε αρκετά στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα, αναρωτιέμαι τι γίνεται, διότι συνεργαζόμαστε με τον ειδικό εισηγητή αυτή του ΟΗΕ για το δικαίωμα για διατροφή και υποχρεωνόμαστε να δούμε περισσότερο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κλιματολογικές αλλαγές είναι ένα θέμα όπου αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι η Φιλανδία θα κάνει κάτι επ' αυτού. Και τέλος, υπάρχει συζήτηση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία αρχίζουμε να πραγματευόμαστε και έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά. Σας ευχαριστώ και θα επανέλθουμε πιο λεπτομερώς σε μια επόμενη ευκαιρία. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και σας ευχαριστώ πολύ κυρία Απνό για τα καλά σας λόγια. Τώρα ο κύριος Τιερή θέλει να μας πει λίγα λόγια σχετικά με τη μελέτη και πώς αυτή συνδυάζεται με τις προτάσεις σας για να ενισχυθεί ε, το θέμα. Θα τα πω γαλλικά για αλλαγή τώρα. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή στην αρχή της συζήτησης είναι ότι ακριβώς κάθισαν με την ηρεμία τους, πράγμα που δεν κάνουμε πολύ συχνά, να σκεφτούν τι θα πει mainstreaming και ποια είναι η μεθοδολογία. Μου άρεσε αυτό που είπε ε, η καθηγήτρια, ότι όταν διαποτίσει ε, όλες τις πολιτικές, η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό είναι το mainstreaming. Και πραγματικά όλοι οι τμήματάρχες, ε, όλοι οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διευθυντές θα πρέπει ακριβώς να ενστερνίζονται ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι οι πρωταγωνιστές, αν το πράξουν αυτό ε, στα διάφορα επίπεδα δράσης, εάν είναι διαποτισμένοι από αυτό το πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε ε, υπάρχει εγγύηση ότι θα τα mainstreamάρουμε καλύτερα και λυπάμαι και για τον νεολογισμό, ζητώ συγγνώμη. Εμείς οι μη κυβερνητικέ οργανώσει το έχουμε θέσει αυτό με κάποιο άλλο τρόπο όταν ζητήσαμε ομάδε εργασία του Συμβουλίου να ασχολούνται περισσότερο με τα κράτη-μέλη. Και όταν ζητούσαμε, που ζητάμε ακόμα να έχουμε πρόσβαση σε αυτέ τι γεωγραφικέ ομάδε, Δηλαδή όχι το COHOM, την επιμέρους επιτροπή, αλλά και για την επιτροπή για την Ασία, για τη Λατινική Αμερική, για άλλα ε, μέρη του κόσμου, για να έχουμε ε, την κατάρτιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για μια γεωγραφική περιοχή της γης. Θα πρέπει λοιπόν έτσι να διαποτίσουν για το πνεύμα των όσων παίρνουν τις αποφάσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο θεματικών ενωτήτων. Τώρα, για το mainstreaming αυτό το περιβόητο δεν θα πρέπει να αποφύγουμε το πραγματικό ζήτημα που είναι η σύγκρουση συμφερόντων και τελικά η πολιτική βούληση. Αν μπορεί κανείς να βρει μια κοινή θέση σε 27 κράτη-μέλη για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν θα μπούμε σήμερα σε αυτό, αλλά να το επιβάλλουμε και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να επιβάλλουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της λαθρομεστανάστευσης και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι υπάρχει κυριαρχία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί όλων των ε, επιμέρους πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε θέματα που έχουν να κάνουν κατά τα άλλα με business ή οικονομική ανάπτυξη να μην έχουμε μια θεωρητική αντίληψη για το mainstreaming. Ε, μιλάμε ότι ε, πρόκειται εδώ για σύγκρουση συμφερόντων και αδυναμία καμιά φορά ε, κάποιων κρατών, εταίρων ή των ίδιων μας των κρατών μελών να βάλουν στην πρώτη γραμμή ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχομαι τώρα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Στο παρελθόν επίσης είχαμε πει ότι Υπάρχει εδώ μια κοινή διπλωματική υπηρεσία στη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό είναι ρίσκο, κίνδυνος και για μας και για το Κοινοβούλιο. Είπε η κυρία Μπενουά Ρομέρ ότι η ιδιαίτερη αποστολή αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να θυμίσει, να θυμίζει την ανάγκη αυτή. Και αυτό είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ε, το καθήκον να εκπροσωπεί το ευρωπαϊκό συμφέρον απέναντι στο καθημερινό, ε, ίσως και ιδιωτελές συμφέρον των κρατών μελών. Δεν θέλω να μειώσω τα κράτη-μέλη, αλλά ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Και αν υπάρξει μια τέτοια υπηρεσία κοινή, ίσως αποδυναμωθεί ο ρόλος των θεσμικών οργάνων και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ασκήσουμε κάποιο αντίβαρο. Συγγνώμη, Πρόεδρος, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θέλω να δώσω το λόγο και στον κύριο Ομπιόλς για να κλείσει. Και, και τελειώνουμε και στις 6.30 κατά τα άλλα, τοπική. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ομπιόλ. Ε, πρόεδρε, εγώ είχα ε, την πρόθεση να προβοκάρω. Έτσι με τρόπο κάπως ε, πιο ευπρεπή να σας προκαλέσω λίγο για να συνεχίσουμε άλλη φορά αυτή τη συζήτηση όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Και νομίζω ότι θα μπορούσε η Πρόεδρος να σκεφτεί ποιος θα ήταν ο κατάλληλος τρόπος ή το σχήμα για να έχουμε ένα τέτοιο διάλογο πιο εμεριστατωμένο και ενδελεχή. Και με το δίκτυο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και για την έκθεση αυτή για το mainstreaming. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να πω σε σχέση με τον όρο mainstreaming ότι αισθάνομαι και εγώ την ίδια δυσφορία με την κυρία Μπενουά Ρομέρ. Όταν είπε ότι δεν υπάρχει μετάφραση αντίστοιχο όρος στα γαλλικά, ούτε στα ισπανικά υπάρχει. Και μου φαίνεται παράλογο να μετράμε πόσες φορές αναφέρεται στις εκθέσεις ο ρόλος mainstreaming σε μια ετήσια έκθεση από χρόνο σε χρόνο. Αυτό το mainstreaming νομίζω θα πρέπει να έχει δύο βασικούς ε, προορισμούς, ε, ε, μάλλον προσανατολισμούς καλύτερα. Όσο γίνεται μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή στην πολιτική και όσο γίνεται μεγαλύτερη πολιτική βούληση προς τα εκεί. Γιατί το mainstreaming είναι θετικό και όλοι συμφωνούμε, αλλά εξαρτάται ε, ουσιαστικά από τη δύναμη ε, του ρεύματος αυτού. Αν θέλουμε αυτό το stream, το ρεύμα να συμπαρασύρει και να ε, συγκεράσει όλες τις πολιτικές της Ένωσης, να έχουμε ένα ρεύμα λοιπόν, αλλά τι να το κάνω το stream αν δεν κινείται. Θα ήταν αρνητικό αν δεν είχε και ροή αυτό και ήταν στάσιμα τα νερά θα πρέπει να βάλουμε εκεί την έμφαση, την πολιτική βούληση, τις δράσεις και τη συνοχή και τη συνέπεια. Και εδώ έχουμε διπλή έννοια, συνέπεια και συνέχεια των διαφόρων ε, θεσμικών οργάνων, αλλά και συνέπεια και συνέχεια όπως είδαμε πρόσφατα ε, μεταξύ συμφερόντων και αξιών γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πέσουμε στη διπλή υποκρισία, να κάνουμε ένα επιμερισμό εργασίας, όπου το Συμβούλιο και μέρη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι οι κακοί που εκπροσωπούν συμφέροντα και το Κοινοβούλιο να είναι ο καλός και να ε, πρεσβεύει και να υπερασπίζει αξίες. Αυτό θα ήταν και υποκριτικό και άκρος αναποτελεσματικό. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε εκεί ένα μέσο όρο, γιατί τελικά οι αξίες για τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες είναι και συμφέροντα. Έτσι, θα πρέπει να υπερασπίζουμε τις αξίες μας με την ίδια ισχύ, το ίδιο στένος και την ίδια ένταση, με αυτό το ίδιο έντονο και ε, ισχυρό ρεύμα που υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Το δεύτερο. Υπάρχει μία λέξη απαγορευμένη από όλες τις εκθέσεις και όλα τα έγγραφα που γράφουμε, που συζητάμε σε αυτή εδώ την Επιτροπή για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ποιο είναι αυτό το ταμπού, απαγορευμένη λέξη, ανύπαρκτη και πουθενά δεν φαίνεται, είναι η λέξη πολιτικά κόμματα. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές, αλλά όταν μιλάμε για διάλογο σε πολιτικό επίπεδο, διαδραστικό και ό,τι άλλο θέλετε, και λέμε ότι θα πρέπει αυτός να γίνεται μεταξύ θεσμικών οργάνων, κοινοβουλίων και εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, λησμονούμε κάτι που μπορεί να είναι ατελές και χωράει ως κριτική θέλετε, που είναι τα βασικά εργαλεία χωρίς τα οποία δεν υπάρχει δημοκρατία και αυτά είναι τα πολιτικά κόμματα. Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών κρατών μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι εφόσον υπάρχουν κοινοβούλια αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτικών κομμάτων. Εντάξει, αλλά αφού συζητούσαμε για την κατάσταση στη Μεσόγειο, τα πολιτικά κόμματα είναι απαγορευμένα ή περιθωριοποιημένα σε πολλά από τα τρίτα κράτη της Μεσογείου και πρέπει να έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στο διαδραστικό πολιτικό διάλογο που με τρόπο πάρα πολύ σωστό και καλό γίνεται. Είναι αυτό που μας είπαν οι πρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές. Πολύ ε, ωραία αυτό που μας είπατε κύριε Μπιόλς. Τώρα, να κάνω εγώ μια πρόταση. Πολλοί από εσά είπατε ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη συζήτηση αυτή και το διάλογο. Είπατε επίσης ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη η συζήτηση και χρειάζεται να συνεχιστεί. Εδώ, σε επίπεδο ε, υποεπιτροπής. να μπορούν να συμμετέχουν και άλλα θεσμικά όργανα, εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων του Ινστιτούτου της Βενετίας και τους ευχαριστώ για την παρουσία και για το γεγονός ότι ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση την τόσο ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Βεβαίως θα γίνουν μεγάλες συζητήσεις σε όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά επανέρχομαι σε αυτό που ήθελα να σας πω στην αρχή. Λοιπόν, αύριο έχουμε δύο πολύ σημαντικές συζητήσεις. Ε, το ένα είναι η Κίνα και η Ουιγούροι. Θα έρθει και η κυρία Γκάλε στις 9 το πρωί. Και στις 10.30 θα ασχοληθούμε με το Ιράν. Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ την κυρία Αρνό και όλους τους υπόλοιπους για τις συζητήσεις και για τις προτάσεις που μας κάνατε.